παρακαλώ να καθίσετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται. Άρχεται η συνεδρίαση. Αν έχει την καλοσύνη παρακαλώ να καθίσετε. Ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο γύρο και για το δεύτερο αυτό γύρο εκλογής του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έλαβα καμία νέα υποψηφιότητα. Εκτός αυτού μου ανακοινώθηκε ότι όλες οι υποψηφιότητες του πρώτου γύρου εξακολουθούν να ισχύουν. Παρακαλώ λοιπόν να μοιράσετε τα ψηφοδέλτια. Γνωρίζετε όλοι σας τη διαδικασία. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, ψηφολέκτες ε, να λάβουν τις ε, θέσεις τους. Οι ψηφολέκτες παραμένουν οι ίδιοι και σας παρακαλώ πολύ να πάτε στις κάλπες για να ψηφίσετε και θα ήθελα να σας παρακαλέσω καταρχήν να απευθύνομαι στους ψηφολέκτες. Κάντε μου ένα μήνυμα αν φτάσετε στις θέσεις σας. Ξέρω ότι στο S, το γράμμα S, για αυτό έχει προβλεφθεί ο κ. Σόκμαρκ, ο οποίο όμω δεν έχει έρθει. Και τον παρακαλώ ή δυνατόν να μεταβείτε στο συντομότερο δυνατόν στο γράμμα S. Και ρωτώ, είναι στη θέση τους όλοι οι ψηφολέκτες. Αλλά από ό,τι βλέπω κανείς δεν μου δίνει σημασία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Φαντάζομαι έχουν έρθει όλοι. Η κυρία Ντότς είναι στη θέση της, ε, είναι οι ψηφολέκτες ε, όλοι στη θέση της. Η κυρία Ντότς συνοδεύεται και από το μωράκι της. ich möchte fragen ob alle abgeordneten ihre stimme abgegeben haben. Μήπως επιθυμεί κάποιος να έχει λίγο περισσότερο χρόνο για να ψηφίσει. Επαναλαμβάνω. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. αν έχετε τελειώσει, παρακαλώ πολύ ε, να μου κάνετε ένα νόημα. Ο συνάδελφος φαντάζομαι θέλει να ψηφίσει. Έχω κάποιες ερωτήσεις, ίσως ε, μπορείτε να με δώσετε λίγη σημασία. Ε, ψηφίσατε παρακαλώ όλοι οι βουλευτές. Ε, αν θέλετε λίγο χρόνο ακόμα, εντάξει, συνεχίζεται η διαδικασία. Για τρίτη φορά. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Μήπως υπάρχει κάποιος στην αίθουσα ο οποίος ε, δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Τότε θεωρώ ότι έληξε ο γύρος αυτός ε, ψηφοφορίας και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μεταβούν στην αίθουσα R11. Η ε, συνεδρίαση διακόπτεται, θα ε, ξαναρχίσει όταν θα ακούσετε το κουδούνι και θα το δείτε και στις οθόνες σας. Προς το